Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε, Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη έχουμε την κοινή συζήτηση για τα χρηματοδοτικά μέσα και μάλιστα έχουμε πολλές εκθέσεις. Πρώτα απ' όλα η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του κυρίου Γκέρενς για το μηχανισμό, μηχανισμό χρηματοδότησης αναπτυξιακής συνεργασίας, μετά σύσταση για δεύτερη ανάγνωση των κυρίων Λόχμπιλ και Γκάλ, χρηματοδοτικό μέσο για την παραγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, κατόπιν σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του κυρίου Μίτσελ, Μηχανισμό χρηματοδότηση αναπτυξιακή συνεργασίας και σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του κυρίου Σόλτ, θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένε χώρες. Πρώτα απ' όλα θα λάβουν το λόγο όλοι οι εισηγητέ και πρώτα απ' όλα ο κύριος Γκέρνς για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Το σχέδιο κανονισμού που συστήνει ένα μηχανισμό με συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα για τις χώρες ΑΚΕ εξετάζεται σε δεύτερη ανάγνωση σήμερα. Σας υπενθυμίζω ότι στην πρώτη ανάγνωση ταχθήκαμε υπέρ ε, των μέτρων που θα βοηθήσουν τις χώρες που εξάγουν μπανάνα διότι ε, λοχεύει ο κίνδυνος να επιδεινωθεί η κατάστασή τους λόγω της σύναψης συμφωνίας των ΠΟΕ με ε, άλλους παραγωγούς από τη ΣΥΠΑ και από τη Λατινική Αμερική ούτως ώστε να επιληθεί η εμπορική διαφορά που σχετίζεται με τους ε, δασμούς για την μπανάνα. Οι εισαγωγικοί δασμοί για την μπανάνα βάσει αυτής της συμφωνίας θα φθήνουν από 176 ευρώ ευρώ ε, τον τόνο 114 ευρώ μέχρι το 2017. Αντίθετα, οι μπανάνες που έρχονται από τις χώρες ΑΚΕ θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ε, ατελή εισαγωγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, θα είναι λιγότερο ευνοϊκή η κατάσταση μετά την ε, θέση σε ισχύ αυτής της συμφωνίας και έτσι άρχισαν οι χώρες ΑΚΕ τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα. Η Επιτροπή Ανάπτυξης, της οποίας είμαι ο εισηγητής, την πρώτη ανάγνωση Ένωση ε, κατάφερε να ε, υποβάλει τροπολογίες που βελτιώνουν το αρχικό κείμενο της συμφωνίας. Επίσης τονίζουμε τη σημασία της εκρίζωσης της στόχης ε, και της αναβάθμισης των συνδικών εργασίας και διαβίωσης που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Οι γεωργοί και οι μικρές επιχειρήσεις επίσης θα πρέπει να θεωρηθούν ως οι βασικοί δικαιούχοι αυτών των μέτρων τρίτων. Ο κανονισμός ε, ε, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιβάλλον, ε, στην υγεία και στους κανόνες εργασίας. Επίσης, χρειαζόμαστε κριτήρια διαφάνειας για την κατανομή των κονδυλίων και προβλέπονται μέσα στη συμφωνία. Επίσης, χρειάζεται 18 μήνες πριν εκπαινεύσει το πρόγραμμα να υπάρξει σχετική κοινοποίηση από τις χώρες ΑΚΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν συμφωνία για τη χρηματοδότηση των συνοδευτικών αυτών μέτρων για την περίοδο 2010-2011. Ε, η πρόοδος που σημειώθηκε καλύπτει τις προσδοκίες ε, των χωρών ΑΚΕ. Το μόνο σημείο ρήξη σχετίζεται με ένα οριζόντιο θέμα, δηλαδή την ε, εφαρμογή των πράξεων κατεξουσιοδότης σε σχέση με την λειτουργία, τη συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το άρθρο 293 αποτελεί την ιδανική νομική βάση για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποφανθεί για τα στρατηγικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής αναπτυξιακής βοήθειας. Μέχρι τούδε το Συμβούλιο δεν αναγνωρίζει ε, τον δέοντα ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη για τη χρηματοδότηση αυτού του μηχανισμού. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι και το τονίζω όλο ιδιαίτερο ότι αρνούμαστε να ε, ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική του Συμβουλίου γιατί δεν οδηγεί ε, σε τίποτα και φαίνεται αυτό από την καθημερινή δράση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Καλό τους ε, συναδέλφους να υποστηρίξουν αυτή τη θέση την οποία καταλήξαμε ε, στην πρώτη ανάγνωση και σας ε, καλώ να υπερψηφίσετε το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο σήμερα σας παρουσιάζω. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λοχμπίλτερ έχει το λόγο και αυτή άλλα τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανάπτυξη δημοκρατικών δομών αλλά και η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι οι βασικές απαιτήσει στην Ιεμένη, στην Τινησία, στην Αίγυπτο, όλων αυτών που κατέβηκαν στους δρόμους ειρηνικά και με την ελπίδα θα επιτύχουν την αλλαγή. Όλοι οι λαοί λοιπόν του Μαγκρέπ και του αραβικού κόσμου διεκδικούν το δικαίωμα για την ελευθερία έκφρασης και ελευθερία τύπου, τη δυνατότητα ελευθέρων εκλογών και πλήρους συμμετοχής στα τεκτενόμενα της χώρας τους. Το εργαλείο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει σαν στόχο να υποστηρίξει αυτά τα δικαιώματα και μέχρι στιγμής έχει μπορέσει να δράσει μονάχα σε περιορισμένο βαθμό στις χώρες αυτές, γιατί στις χώρες αυτές είναι γεγονός ότι όλοι αυτοί που έχουν διαφορετική άποψη από την επικρατούσα της κυβέρνησης είναι αντικείμενο καταδίωξης έχουμε συντάξει σχέδια συγκεκριμένα για καλύτερη χρησιμοποίηση αυτών των ε, κονδυλίων, επομένως με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη δημοκρατία. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία αυτή στην Τινησία. Θα ήταν πολύ θετικό από αυτές τις ενέργειες να προκύψει ένα μελλοντικό υπόδειγμα το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες χώρες της περιοχής ώστε να υπάρξει μια γενική και συνολική ε, μεταλλαγή. Η Κομισιόν ε, έχει αναγνωρίσει τη σημασία και της ε, αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πηγαίνει στην Τινησία και που θέλει να υποστηρίξει θέματα όπως η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να υποστηρίξουμε όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία στις χώρες αυτές. Μπορούν να είναι κυβερνητικοί φορείς, μπορούν να είναι ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, Ινστιτούτα πολιτικού χαρακτήρα, μπορούν να είναι μεμονωμένα άτομα. Έχουμε λοιπόν μία δομή η οποία νομίζω ότι μας επιτρέπει κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ακόμα και χωρίς την έγκριση των τοπικών κυβερνήσεων. Αυτό δεν αποτελεί μια <clears throat> ανάμειξη στα εσωτερικά του θέματα, γιατί η φύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τέτοια που δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την κρατική πίεση και βία και θα πρέπει να ισχύει σε οικουμενικό επίπεδο. Προφανώς θα πρέπει εμείς όλα αυτά τα σχέδια και την στοχοθεσία της, ε, των εργαλείων για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα έχουμε υπό συνεχή εξέταση και επισκόπηση μέχρι ε, μέχρι στιγμής αυτά τα εργαλεία ήταν σχετικά καινοφανή και δεν ήταν δυνατό να έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση της επίπτωσής τους. Αυτό το οποίο κάνει ακόμα πιο σημαντικό να μπορέσουμε να προβούμε σε καλύτερες ε, ε αξιολογήσεις στο μέλλον. Αυτά θα πρέπει να έχουν το στόχο να διασαφηνίσουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων και των μέσων και να μπορέσει να καθορίσει με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση μια καλύτερη στοχοθεσία στα θέματα αυτά. Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε <clears throat> πάντα διαπιστώσει ότι με μικρές χρηματοδοτικές ικανότητες μπορούμε να αρρωγήσουμε σχέδια τα οποία παίζουν ένα σημαντικό ρόλο μέσα σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο και τίθεται επίση και το θέμα αυτό στα πλαίσια του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δεχτούμε να υπάρξει μια περικοπή της χρηματοδότησης αυτών των σχετικά ε, περιορισμένων εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εξουσιοδότηση πράξης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε τομείς όπως οι μεταφορές και το περιβάλλον δεν υπάρχει καμία διαφωνία σε σχέση με τις κατεξισοδότηση πράξεις. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ επίμαχο θέμα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Αλλά αμέσω μετά από την έγκριση της ε, Συνδίκης Λισαβόνας είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματά του στην απόφαση μέσα στα στρατηγικά προγράμματα για την χρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων στις ε, χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λόχ Μπίλτερ. Η κυρία Γκάλ και αυτή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, όλα όσα είπε μόλις η κυρία η αγαπητή συνεισηγήτρια, έχουν πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα, ειδικά αν σκεφτούμε το ότι αυτή τη στιγμή οι διεθνείς κατάσταση είναι τεταμένη. Είχαμε χθε συζήτηση περί Αιγύπτου και την Ισία και αυτό μας δείχνει πως ε, πρέπει να δείξουμε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το <laughs> μηχανισμό χρηματοδότησης ε, για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων ε, του ανθρώπου. Είναι ένας σημαντικός λόγος αυτός για το να έχει το Κοινοβούλιο πλήρη δικαιώματα κοινοβουλευτικού ελέγχου αυτών των ε, μέσων. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε κοιτάξαμε ζητήματα ουσίας τα οποία αφορούσαν ε, το πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τοπικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λειτουργήσουν σωστά. Εδώ πέρα κοιτάμε την άλλη πλευρά του νομίσματος στη δεύτερη ανάγνωση. Μιλάμε για τα δημοκρατικά προνόμια που έχει το Κοινοβούλιο στο θεσμικό πλαίσιο. Κοιτάμε λοιπόν αυτούς τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, ειδικά της δημοκρατίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου και εδώ πέρα έχουμε μία πάλι μεταξύ των θεσμικών οργάνων γιατί με τη συνθήκη της Λισαβόνας και της πράξης κατεξιοδότηση παραδείγματος χάρη έχουμε περισσότερες εξουσίες και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δημοκρατικά δικαιώματά μας γιατί όπως σας είπα μιλάμε για πράξεις κατά εξουσιοδότηση και έχουμε το πρώτο σαφές παράδειγμα του ρόλου, ε, της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου. Οπότε πιθανότατα στην ε, διαδικασία της ε, συνδιαλλαγής ε, εμείς δηλαδή το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας για κοινοβουλευτικό έλεγχο και φαντάζομαι πως ε, με τους ε, συνεισηγητές ε, θα συμφωνήσουμε πως πρόκειται για κάτι το οποίο έχει εξαιρετική σημασία. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κράτος δικαίου προστατεύει τη δημοκρατία. Αυτό είναι το νόημα εδώ πέρα της Θέλουμε να βοηθήσουμε γυναικόπαιδα να εκμεταλλευτούν πλήρως τα δικαιώματά τους, ανθρώπους οι οποίοι ε, αγωνίζονται κατά των βασανιστήριων. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη θανατική ποινή, θέλουμε να βοηθήσουμε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συνεχίσουν να κάνουν το ζωτικό τους έργο. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε οι δικαιούχοι εδώ πέρα, δηλαδή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παλεύουν σε πολύ δύσκολες ε, συνθήκες να λάβουν τη βοήθεια που τους ε, αξίζει. Γι' αυτό ακριβώς εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να έχουμε λόγο στη δημιουργία αυτών των στρατηγικών προγραμμάτων πλαισίου. Και όταν ε, μιλάμε για μελλοντικά σχέδια πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε λόγο και επίσης αντιλαμβάνομαι πως θα ε, γίνουν ακόμη σημαντικότερα βήματα και θυμάστε την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μας είχαν ζητήσει γνωμοδότηση. Όταν μιλάμε λοιπόν πως έχουμε περάσει σε μια εποχή μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας θέλουμε να λειτουργήσουμε και με ανάλογο πνεύμα και ελπίζουμε Κομισιόν και Συμβούλιο να αναγνωρίσουν τη σημασία αυτών στην διαδικασία συνδιαλλαγής. Ευχαριστώ κυρία Γκάλ. Ο επόμενος εισηγητής είναι ο κύριος Σόλτς, επίσης για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το χρηματοδοτικό μέσο για συνεργασία με τις ε, εκβιομηχανοποιημένες χώρες ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να διαθέσουμε άνω των 300 εκατομμυρίων για ακαδημαϊκή συνεργασία, Erasmus Mundus, ε, πολιτιστική συνεργασία και ευημερή σχέση. Ειδικά επίσης θα ληφθούν υπόψη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης ε, με το λεγόμενο ICI είναι το ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, έργα σε αναψώμενες χώρες, μάλιστα έργα τα οποία δεν εμπίπτουν στο γενικότερο ορισμό της αναπτυξιακής βοήθειας, όπως παραδείγματος χάρη αποστολή Ευρωπαίων φοιτητών σε πανεπιστήμια της Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής. Ακριβώς οι νέες ε, αυξημένες ευθένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα αναπτυσσόμενα κράτη ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Με την αναδιατύπωση λοιπόν του κανονισμού έχουμε αναλάβει αυτή την εργασία για να μπορέσουμε να αποκριθούμε στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Ορίζεται λοιπόν σαφώς ποιος ε, μπορεί να λάβει χρηματοδοτική στήριξη και με ποιες ε, προϋποθέσεις και για ποιο σκοπό. Θα πρέπει επίση να φροντίσουμε οι χώρες αυτές τηρούν τις βασικές διατάξεις για την προστασία της εργασίας και να υπάρξει και μια σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου για να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή. Επίσης, ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριληφθούν σε αυτή την συνεργασία. Θα ήθελα επίσης να τονίσω πως θεωρώ απολύτως απαραίτητο να τηρήσουμε τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην γίνει καμία παραχώρηση ως προς αυτό. Όταν μιλάμε για χρηματοδότηση αναψηφωμένων χωρών θα πρέπει να δούμε την συνοχή της πολιτικής ειδικά όσον αφορά τα μέτρα καταπολέμησης της κρίσης τροφίμων. Στην πρώτη ανάγνωση αποφασίσαμε κατά πλειοψηφία, έστω και με μικρή πλειοψηφία, να μην ε, δώσουμε χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε πως πηγαίνουμε στην ε, δεύτερη ανάγνωση με μια επιταχυμένη διαδικασία. Το ICI Plus θα πρέπει να προσαρμοστεί με, από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις νέες απαιτήσεις και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής ε, όλα πάνε καλά από αυτά τα οποία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια. Αλλά βλέπετε πως ε, η κατανομή των αρμοδιοτήτων που ορίζεται στην συνθήκη της Λισαβόνας ε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδειχθεί σε αυτόν τον τομέα. Μιλάμε για το ζήτημα της δημοκρατίας με τις πράξεις ε, κατεξιοδότηση. Οπότε Κομισιόν και Κοινοβούλιο έχουν και τηρούν δυστυχώς διαφορετική άποψη από το Κοινοβούλιο. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν. Εμείς θέλουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι των ψηφοφόρων μας. Θέλουμε αποδείξεις για την εφαρμογή των ε, πολιετών σχεδίων Κομισιών και Συμβουλίου σύμφωνα με το κοινοτικό πνεύμα. Από τη συνδίκη Ιδέα της Λισαβόνας ο νέος μας ρόλος είναι υποχρέωση του νομοθέτη και θέλουμε δικαίωμα βέτο όλα τα μέτρα χρηματοδότησης της ε, εξωτερικής πολιτικής, εδώ πέρα συμφωνούν ε, και οι πρόεδροι της ομάδας και της Επιτροπής, θα πρέπει να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτά τα οποία συμβαίνουν ε, και η συμπεριφορά που έχει επιδειχθεί σημαίνει πω αυτή η αρχή δεν γίνεται ακόμη σεβαστή από τα τρία θεσμικά όργανα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτούμε να έχουμε δικαίωμα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο γιατί η Κομισιόν θα πρέπει να υπόκειται στη θέληση του νομοθέτη και όχι στη αυτά τα οποία ορίζει σαν ανακοινώσει. τη. Σας ευχαριστώ. Επειδή ο κύριο Μίτσελ δεν είναι ακόμα εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ντεχούχτα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Αντικαθιστώ τον Αντρέ Σπίλμπαγκ. Είναι στην Αλοδαπή, είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις ε, και τον αντικαθιστώ εγώ στη σημερινή συζήτηση για τις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή συνεργασία. Ευχαριστώ όλους τους συγητές, ε, την κυρία Γκάρελ, την κυρία Λόχ Μπίλερ, τον κύριο Μίτσελ, ε, τον κύριο Σόλτς και τον κύριο Σάλ Γκέρενς. Έχουμε, είχαμε μια αγαστή συνεργασία και πέρα από τις πράξεις κατεξουσιοδότηση υπάρχει ευρεία συνένεση ανάμεσα στα συναρμόδια θεσμικά όργανα. Ε, εκρεμούν ε, κάποια ζητήματα ακόμη λόγω ε, της διαμόρφωσης της νέας διοργανικής σχέσης, το νέο περιβάλλον με τη νέα συνθήκη. Ε, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή από πολιτικής και οικονομικής πλευράς ε, και ε, δεν κατανοούν κάποιοι ότι η εφαρμογή αυτών των πράξεων ε, είναι ένα εσωτερικό θέμα, θέμα εσωτερικής κατανάλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Πάντω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με τους στόχους Ευρωπαϊκή Πολιτική ε, στον τομέα του εμπορίου ε, και το ίδιο και για τι εξωτερικέ σχέσει. Από την τελευταία συζήτηση που έγινε τον Οκτώβρη καταλήξαμε στη συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβάλλει το άρθρο 293 όπου προβλέπεται η επωνομαζόμενη διαδικασία της πράξης κατεξουσιοδότηση που θα χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων και των πολιετών σχεδίων δράση. Ε, ο Συμβούλιο όμω απόρριψε τι σχετικέ τροπολογίε ε, του Κοινοβουλίου ε, στην πρώτη ανάγνωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία κυρίω για το ΑΚΕΣΥΝ και για την, την πρόταση για τα συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες. Ουδάλλως δεν δίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτελέσει το σχετικό τμήμα του προπολογισμού. Ειδικότερα για το ΑΚΕΣΥΝ... Ε, συμφωνούμε ότι το εργαλείο αυτό θα προαγάγει τις σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τις εκβιομηχανισμένες ε, χώρες και πρέπει να είμαστε ε, διοικητικά έτοιμοι για την εφαρμογή αυτών των πράξεων. Μιλάμε επίσης για την ενεργειακή συνεργασία, υποστήριξη επιχειρήσεων, στόχους περιψηφιακού θεματολογίου και ούτω καθεξής. Συγκεκριμένα για τα συνοδευτικά μέτρα της μπανάνας μπορώ να τονίσω και ελπίζω να έχει απήχηση αυτό που λέω ότι όλα αυτά τα ζητήματα συνδέονται αλληλένδετα με τη Συμφωνία της Γενέβης ε, που θέτει πέρασε σε μια μακρά ε, αντιδικία που είχαμε στον ΠΟΕ και στον ΚΑΤ. Εδώ και 20 χρόνια περίπου διαρκεί αυτή η εμπορική διαφορά και θα στηρίξουμε 10 χώρες εξαγωγής μπανάνας, ε, χώρες ΑΚΕ. Θα μειωθεί δηλαδή το προτιμησιακό περιθώριό τους που προκύπτει από τις συμφωνίες της Γενέβης. Είναι εξόχως σημαντικό το θέμα γιατί ε, διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ήδη ε, ε, κυρίως ενώπιον των παραγωγών χωρών ΑΚΕ. Ε, σε σχέση τώρα με την επιζητιστική ασφάλεια και τα δεινά που υφίσταται διάφορες χώρες αντιλαμβανόμαστε πόσο κάποια κράτη εξαρτώνται αποκλειστικά από την εισαγωγή κάποιων βασικών αγαθών. Είναι κατεπήγον το θέμα, το αντιλαμβάνεστε. Ε, και καταλαβαίνω και την ανησυχία του Κοινοβουλίου γιατί εμπλέκεται στο στρατηγικό σχέδιο και στην εκπόνηση των πολιετών σχεδίων δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει εισηγήσεις για να ενισχύσει τον έλεγχο από πλευράς του Κοινοβουλίου και ε, ότι πρότεινε άλλε συμβαστικέ λύσει. Ε, πλην όμως ε, δεν έγιναν αποδεκτές ε, και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να τονίσω τώρα τη δέσμευση που ανέλαβε τον περασμένο Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέβριση πολιτικών λύσεων. Τα τρία θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή, θα πρέπει να συμφωνήσουν κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάγνωσης, ούτω ώστε να υλοποιήσουν τη δέσμευσή του και να, κατόπιν να υλοποιήσουν το σχέδιο αυτό. Είναι δημοσιονομικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό το θέμα και θα έχει σοβαρέ συνέπειε. Ταυτόχρονα, εφόσον ε, τροποποιήθηκε η Επιτροπολογία με την Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αποδόθηκαν νέε αρμοδιότητε στο Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρότερο ρόλο και νέε υποδομέ, ώστε να εφαρμόζει πιο συνεκτικά ε, και ολοκληρωμένα την εμπορική πολιτική, εξυπηρετώντα του κοινού στόχου. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και αναμένω τι παρεμβάσει σα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε πίτρο. Ερχόμαστε τώρα στους ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Και καταρχήν εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Πόγκα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα θα λάβει θέση για δεύτερη φορά στην, σε σχέση με την τροποποίηση του εργαλείου για την ανάπτυξη και συνεργασία που προβλέπει την εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης στον τομέα της μπανάνας, συνοδευτικών μέτρων. Τα συνοδευτικά αυτά μέτρα οφείλονται στη μείωση των δασμολογικών προτιμήσεων που είχαν δοθεί στις χώρες ε, ΑΚΕ μετά από τη Συμφωνία της Γενέβης το 2009 με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που έλαβε χώρα στη Γενέβη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει με 190 εκατομμύρια τις χώρες εκεί για να αντιμετωπίσουν τη νέα αυτή μορφή ανταγωνισμού. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τροποποιήσει εμείς την πρόταση της Κομισιόν και στην ουσία και σε ό,τι αφορά τον τύπο. Για την ουσία το Συμβούλιο δεν μας ακολούθησε και σήμερα περνάμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοθετήματος αυτού, διότι το Συμβούλιο δεν δέχτηκε την διαδικασία κατ' εξουσιοδότηση να εφαρμοστεί στην στρατηγική και τα ενδεικτικά πολιετή προγράμματα. Και έτσι δεν δέχεται να λάβει υπόψη την πρόοδο της ε, συνθήκης της Λισαβόνας για τα θέματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντιδράσει λοιπόν, πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στις χώρες ΑΚΕ. Έχουμε ήδη κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε τα 190 αυτά εκατομμύρια να απελευθερωθούν και να εκταμιευθούν. Θέλουμε να δώσουμε όμως και ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προασπίσει τα δικαιώματά του όπως αναφέρονται στην ΣΛΕΕ, στην Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λισαβόνα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση ενώδη των χωρών ΑΚΕ και πρέπει το Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του όπως έχει ήδη πράξει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πόγκα. Υπάρχει μια μπλε κάρτα κύριε Πόγκα. Επιτρέπετε να σας θέσει το ερώτημα ο αξιότιμος κύριος βουλευτής. Έχετε το λόγο. Αναρωτιέμαι, αν έχει σκεφτεί κάποτε ο μιλητής ότι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος και ιδίως ο Βρετανός φορολογούμενος μήπως προτιμάει αυτά τα 190 εκατομμύρια να παγώσουν, να μείνουν στην κατάψυξη για πάντα στο δίνεκες. Το έχετε σκεφτεί ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχετε... Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες, μόνο αυτό θα σας θυμίσω, που προβλέπουν δεσμεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις της με τις χώρες ΑΚΕ. Και σε... Ε, θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις της, τις συμφωνίες, οπότε ποτέ δεν το σκέφτηκα ότι θα μπορούσατε να ζητήσετε πάγωμα των 190 εκατομμυρίων. Σας ευχαριστούμε. Προχωρούμε. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τους ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Τυρολιέν. Για ένα λεπτό επίσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κοινώ εκπεφρασμένη θέση ε, η κοινώ εκπεφρασμένη θέση του Κοινοβουλίου καταδεικνύει σε ποιο βαθμό οι αρμοδιότητε εκτέλεση έχουν ε, κέρια σημασία για το σώμα μα. Όμω για τα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα ε, δημιουργείται μία μηχανία ενώπιον των ε, χωρών παραγωγών μπανάνα. Γιατί έχει νομιμοποιηθεί η αντιστάθμιση που έχουν αποκτήσει βάσει των συμφωνίων. Παρόλα αυτά δεν έχουν εκταμιευτεί τα κονδύλια ενώ το προβλέπουν οι συμφωνίε τη Γενέβη. Και γι' αυτό και πάλι σήμερα σήμερα εδώ. Σας απευθύνω έκκληση για την εκτέλεση των συμφωνιών να τηρηθούν ε, τα υπεσχημένα. Το διεκδικούμε διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποφανθεί για την εξωτερική αναπτυξιακή βοήθεια και τι εξωτερικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην πέσουμε στην παγίδα τη Επιτροπή ε, και ε, του Συμβουλίου. Πρέπει να επικρατήσει το πνεύμα τη συνθήκη και εξάλλου αυτό επιτάσσει και επιτάσσουν τα ιστορικά μα βιώματα. Ο κύριο Λάμστορφ δεν είναι εδώ. Οπότε για τους Ευρωπαίους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Ντέβα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ ευγενικό από μέρους σας να μου δώσετε το λόγο νωρίτερα. Το θέμα αυτό έχει τεχνικές πτυχές και ανθρώπινες πτυχές στην πλευρά της φτώχειας. Οπότε είναι κοινή συζήτηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω στο Συμβούλιο πως το Κοινοβούλιο αυτό θα ελέγχει και θα κοιτάει με διαφάνεια και λογοδοσία το πώς ξοδεύουμε τα λεφτά των φορολογουμένων μας όσον αφορά την διεθνή ανάπτυξη. Εάν δεν μπορεί να το αναγνωρίσει αυτό το Συμβούλιο και να αναγνωρίσει πως οι πράξεις κατά εξοδότηση πρέπει να πάνε στο Κοινοβούλιο για να έχουμε δικαίωμα ελέγχου, τότε τι στο καλό κάνουμε εδώ μέσα, κυρία Πρόεδρε. Τι διαβεβαιώσει μπορούμε να δώσουμε στους φορολογούμενους για τα χρήματα που μας δίνουν καλή την πίστη για να ξοδέψει η Κομισιόν στην διεθνή ανάπτυξη. Δεύτερον, για το ζήτημα της μπανάνας, το οποίο επίσης πρέπει να εξετάσουμε. Έχει χάσει και από τις δύο πλευρές ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Είχαμε μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου η οποία έχει αποτύχει και τώρα πρέπει να αποζημιώσουμε τις χώρες που παράγουν μπανάνα και παίρνει το μικρόφωνο του μιλητή η πρόεδρος. Συνεχίζουμε η κυρία Βερζιά. Δεν είναι εδώ οπότε για την Ευρώπη της ελευθερίας και της ε, δημοκρατίας, ο Κόμις του Ντάρτμαθ. Υπάρχει μια δικαιολογία η οποία φαίνεται κάπως αξιόπιστη για κάθε ένα από τα τέσσερα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία εξετάζει σήμερα το Κοινοβούλιο. Αλλά άμα τα πάρουμε ομού και τα τέσσερα, ο στόχος τους είναι να προωθήσουν μια ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Το έκανε σαφές ο κύριο Επίτροπος με την συνηθισμένη του σαφήνεια και ειλικρίνεια και θέλω να τον ευχαριστήσω. Ξέρουμε τώρα ποιο θα πληρώσει την ύφη για όλα αυτά. Ο ξεζουμισμένος φορολογούμενος, όπως πάντα. Και δυσανάλογα ο Βρετανός φορολογούμενος. Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων μου λοιπόν χθε και σήμερα το πρωί εξακολουθεί να είναι άγνωστο το κόστο αυτών των ενεργειών. Η Κομισιόν και πάλι είναι σπάταλη και είναι ανεύθυνη αλλά με λεφτά που δεν είναι δικά τη. Γι' αυτό εμεί δεν υποστηρίζουμε καμία από αυτέ τι προτάσει. Σα ευχαριστώ και για σας υπάρχει μία μπλε κάρτα. Θέλετε να, μπορείτε να απαντήσετε. Βεβαίως. Παρακαλώ κύριε Λάκτφριντ. 30 δευτερόλεπτα. Άψα εδώ πέρα, κύριε Πώς πάντα μιλάτε για το Βρετανό φορολογούμενο. Θα με ενδιέφερε. Θεωρείτε πως εκπροσωπείτε μόνο μία μικρή ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ή θεωρείτε πως εκπροσωπείτε κάπου και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 30 um, uh, um, δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν μπορώ να απαντήσω ανέφερα και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και τον Βρετανό φορολογούμενο στην ομιλία μου. Αλλά εξελέγην από Βρετανούς, από κανέναν άλλον. Οπότε βασική μου ευθύνη είναι βεβαίως έναντι του Βρετανού φορολογούμενου. Αλλά συμπάσχω και με τον δοκιμαζόμενο Ευρωπαίο φορολογούμενο σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και στη δική σας, την Αυστρία η οποία συνεισφέρει και άρα και τα δικά σας λεφτά σπαταλιώνται στην κατασκευή αυτών των ματαιόδοξων και έφραυστων αυτοκρατοριών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Μπράντ εξονόματος των Πρασίνων για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να αντιμετωπίσω μια σειρά από θέματα. Πρώτα απ' όλα να θίξω το θέμα της ευκαμψίας στα χρηματοδοτικά εργαλεία στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι στις ε, πρόσφατες εβδομάδες και πρόσφατες μήνες δούμε ότι υπάρχουν πολλά απρόβλεπτα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο διεθνή στίβο και δεν έχουμε <clears throat> ουσιαστικά καθόλου χρήματα διαθέσιμα για να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει όμως ένα εργαλείο το οποίο είναι ιδιαίτερα πρόσφορο, είναι το εργαλείο σταθερότητας και το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για άλλους στόχους από αυτού του οποίου εκλήθη να εξυπηρετήσει. Καταρχήν, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη λοιπόν ευκαμψία στα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής και αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι αυτό μπορεί να συμβαδίσει μονάχα με αυξημένη δημοκρατική ε, λογοδοσία από την πλευρά της Κομισιόν. Θέλουμε λοιπόν στο μέλλον, εάν χρειάζεται μεγαλύτερη ευκαμψία για τα εργαλεία αυτά, να εξασφαλίσουμε ακριβώς ότι θα υπάρχει αυτή η λογοδοσία δημοκρατική. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε μαζί με τα άλλα κράτη τα οποία ε, ασχολούνται στα θέματα ανάπτυξης συνεργασίας. τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν και πάλι ποια ήταν η σύνδεση της δημοκρατίας και των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε ότι αυτά τα στα κράτη ε, βλέπουν να υπάρχει πολλές φορές συνεργασία εκεί του ΟΗΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να έχουμε καλύτερη συνεργασία μαζί με τον ΟΗΕ. Και εξάλλου τα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική μα κατέδειξαν τη σημασία τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για μένα επίση του θέματο ισότητα των φύλων και πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί στα θέματα αυτά όταν θέλουμε να έχουμε πρόσφορε δομέ για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπράντνερ για του μη εγγεγραμμένου δεν βλέπω τον ομιλητή τον κύριο Γκρίφιν. Ακολουθούμε τώρα με τους υπόλοιπους ομιλητές και δίνω το λόγο στον κύριο Μπρόκ για ένα μισή λεπτό. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να είναι σαφές ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να υπάρχει η διάκριση μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Δεν πρόκειται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει διαχειριστικές αρμοδιότητες ή να αναλάβει την εκτέλεση αυτών των ε, προγραμμάτων. Αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε μια επιταγή εν λευκό στην Κομισιόν για να εκτελέσει αυτά τα προγράμματα. Ιδίω όταν αυτό κινδυνεύει να γίνει κατά της θελήσεως του νομοθέτη. Η κατεξουσιοδότηση πράξεις μας δίνουν πάντα τη δυνατότητα να αναστείλουμε και να ανακαλέσουμε την εξουσιοδότηση αυτή εάν θεωρήσουμε ότι η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών δεν γίνεται βάσει των αρχικών, της αρχικής θέλησης των, του νομοθέτη. Πιστεύουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να δράσουν με ένα πιο λογικό τρόπο ώστε να χάνουμε περισσότερο χρόνο σε τέτοια θέματα εκτέλεσης και επιτροπολογίας. Ε, το Κοινοβούλιο έχει καταφέρει μετά από πολλές προσπάθειες να υπάρχει το εργαλείο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών και τις δημοκρατικές δυνάμεις σε χώρες όπου επικρατεί δημοκρατία. Και βλέπουμε τώρα ότι αντίθετα με τη θέληση του νομοθέτη η Κομισιόν δεν χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα στη Βόρεια Αφρική. Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα. Γι' αυτό, για να τηρηθεί λοιπόν η θέληση του νομοθέτη, θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες για αυτά τα εργαλεία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμισ. Ένα, ένα λεπτό να βγει ε, έξω στον δρόμο, να φύγει ο Μουμπάρακ. Έτσι φωνάζουν στους δρόμους. Με τις διαδηλώσεις στην Αίγυπτο, στην Τινησία και σε άλλες αραβικές χώρες, εκατομμύρια χύνονται στους δρόμους για να καταπολεμήσουν την καταστολή και την διαφθορά, να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για οικουμενικά δικαιώματα. Επαναλαμβάνεται η ιστορία γιατί όλοι υποστηρίζουν τη δημοκρατία για να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, έχει τη δυνατότητα και πρέπει να δράσει για να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φίλων, το κράτο δικαίου, τι ελεύθερε εκλογέ και τη δημοκρατία. Και γι' αυτό πρέπει να είναι τους, ε, τις ενισχύσουμε αυτέ τι χώρε χρηματοδοτικά. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη πολιτική και να χρησιμοποιούμε τα μέσα συνεργασία που έχουμε για την επιδίωξη αυτών των στόχων. και όλα αυτά υπό τον έλεγχο υπό τον, του Κοινοβουλίου και γι' αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή τη διαδικασία των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Ευχαριστούμε κυρία Ευχαριστώ. Ε, ναι, για ένα λεπτό κύριε Μικαλής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχει δίκαιο η κυρία Γκόμες και η κυρία Λοχμπίλερ όταν λένε πως τα γεγονότα στην Αίγυπτο και στην ε, την θα έπρεπε να έχουν τη στήριξή μας και θα έπρεπε να έχουν τραβήξει την προσοχή μας. Πράγματι τα μέσα τα οποία συζητάμε σήμερα μας δίνουν τέτοιες δυνατότητες, ειδικά το χρηματοδοτικό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και είμαι πεπισμένος πως πρέπει να τα υποστηρίξουμε γιατί τα δικαιώματα αυτά είναι παγκόσμια το δικαίωμα να ζει κανείς σε δημοκρατία, το δικαίωμα να ζει σε μια χώρα που αποδέχεται τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι το φυσικό. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι πως το δεύτερο μέσο μας δίνει την δυνατότητα να δίσουμε βοήθεια ανεξαρτήτως του τι θέλουν οι αρχές της εν λόγω χώρας. Και αυτό είναι σημαντικό. Η Ουκρανία χρειάζεται τη βοήθειά μας, πολλές χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και πρέπει να το εφαρμόσουμε και σε αυτές τις χώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ταβάρες για ένα λεπτό. Συζητούμε εδώ μια σειρά από ε, ε δοτικών εργαλείων, όπως αναφέρεται και στην έκθεση του κ. Γκέρνς για την ανάπτυξη, επίσης και στην έκθεση του κ. Σόλτς και άλλων. Είναι πολύ σημαντικό με τα μέτρα αυτά να βελτιώσουμε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και να βελτιώσουμε ακόμα και την νομοθετική πρακτική. Αλλά το Συμβούλιο δεν θέλει να συμπληρώσει τη διαδικασία συναπόφασης που εμπεριέχεται σε αυτά τα εργαλεία. Όταν λέμε συναπόφαση σημαίνει ότι πρέπει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία. Τίποτα δεν δικαιολογεί λοιπόν τη στάση του Συμβουλίου το οποίο προσπαθεί με το δικό του τρόπο να εφαρμόσει το άρθρο 290 της Συνθήκης της Λισαβόνας και να το ερμηνεύσει κατά τα δοκούντα. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή πολλών ατόμων Έχουμε δει τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν με τους πρόσφυγες, μας εμποδίζει να λειτουργήσουν σωστά τους κατα... οι καταβλισμοί των ε, προσφύγων και να έχουμε τη σωστή χρηματοδότηση. Πρέπει το Συμβούλιο να καταλάβει και αυτή τη στιγμή τι θέλετε να αμφιβόλω οι ζωές ανθρώπων και είναι καιρό να αναλάβει τις ευθύνες του και να αφήσει αυτή τη διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Στοιάνοφ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώ ε, θα υποστηρίξουμε όλη τη θέση του Κοινοβουλίου γιατί το Κοινοβούλιο οφείλει να προβάλλει τι νέε αρμοδιότητε που του προσδίδει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Ε, ταυτόχρονα όμω, οφείλουμε να διευρύνουμε και τον έλεγχο ε, που ασκείται από το Κοινοβούλιο και για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση που είναι το αντικείμενο τη σημερινή μα συζήτηση. Χρειάζεται και υστερόχρονο έλεγχος μετά την εκταμείευση των κονδυλίων γιατί εκατομμύρια ευρώ απορροφούνται μέσα από αυτά τα προγράμματα και μπαίνουν δυστυχώς στις τσέπες ε, δικτατόρων ενώ στις χώρες μας ε, ε, υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια άποροι. Ε, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι χρησιμοποιούμε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιβιώνουν οι δικτάτορες και όχι μόνο επιβιώνουν, να ζουν πολυτελώς ε, και προσπαθούν ε, να μας ε, ρίξουν καπνό μπροστά στα μάτια για να μην βλέπουμε. Χρειάζεται εξονυχιστικό έλεγχος. Ευχαριστούμε η κυρία Ματέρα τώρα για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, για μια ακόμα φορά να δράσουμε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσουμε τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθαγιάζονται από την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 όπως και στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής μας, των κοινωνικών θεμάτων και της εξωτερικής μας πολιτικής. Ο κανονισμός 1889 του 2006, ο οποίος θεσπίζει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την προώθηση τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο είναι και ευέλικτο και μπορεί να αντιμετωπίσει τις έκτατες καταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Οι συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον αγώνα για τον πολιτισμό μέσα από στρατηγικές συνεργασίας και σωστή δράση των εργαλείων αυτών σε χρηματοοικοδοτικό επίπεδο, η ακόμα περισσότερη μεγαλύτερη ορατότητα και αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να έχει ένα υπεύθυνο χαρακτήρα και τον κοινοβουλευτικό δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω όλες τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατεθεί, οι οποίες ακολουθούν αυτήν την αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις. Ähm, ευχαριστώ. πάρα πολύ. Κυρία Ματέρα, υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Μιγκάλσκι. Το δέχεστε? Δέχεστε την ερώτηση. Παρακαλώ. Κύριε Μιγκάλσκι, έχετε μισό λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να μας πει η κυρία Ματέρα εάν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα ήθελε να δώσει ειδική στήριξη από Πλευρά δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, Λευκορωσία και άλλες χώρες της Ανατολικής Εταιρική σχέση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Πράγματι ναι, η ομάδα μου, το ΕΛΚ, κάθε μέρα αγωνίζεται για αυτό το στόχο, ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο να τύχουν σεβασμό. Εγώ νομίζω ότι οι παρεμβάσει των εξεχών, των συναδέλφων που έλαβαν προηγουμένω το λόγο έχουν επιβεβαιώσει και έχουν υποστηρίξει απόλυτα την πολιτική αυτού του Κοινοβουλίου και εγώ θέλω και πάλι να υπογραμμίσω το γεγονό ότι είμαι σε μια πολιτική ομάδα, το ΕΛΚ, που είναι πεπισμένοι ευρωπαϊστέ, σίγουροι ότι η δράση αυτό το, Ευρω... το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έχει μεγάλη σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρο. Ακολουθούμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Χάουιτ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι σε σχέση με την κοινοβουλευτική εποπτεία και στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τη διαθρωμένη συνεργασία με την οποία είχαμε. Πρέπει να υπάρχει φυσικά και ένα βαθμό εμπιστευτικότητα μερικέ φορέ στα θέματα τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη υποστήριξή του και έτσι πρέπει να συνεχίσει και στο μέλλον. Θέλουμε να έχουμε σχέδια τα οποία θα είναι υψηλή ποιότητα. Πρέπει όμω να μην είναι απλώ κατακαιρματισμένα, αλλά να υπάρχει και μια ολοκλήρωσή του και ελπίζω ότι η νέα υπηρεσία εξωτερική δράση θα μα δώσει τη δυνατότητα να συντονίσουμε καλύτερα αυτά τα προγράμματα. Ελπίζω θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και θέλω να εξασφαλίσω ότι κάποια από αυτά τα προγράμματα πράγματα τα οποία αυτή, τη στιγμή προετοιμάζονται χρειάζεται να έχουν αρρωγή σε νομικό επίπεδο από άτομα με υψηλά προσόντα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αίγυπτο και σε άλλα μέρη στον κόσμο ξέρουμε ότι θα ζητήσουν ακόμα περισσότερη χρηματοδότηση για δράση υπέρ τη δημοκρατία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη παρακολούθηση των εκλογών. Θέλουμε να παραμείνει λοιπόν ένα σταθερό ποσοστό μέσα σε αυτόν τον κανονισμό για τα προγράμματα αυτά ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά χρειαζόμαστε και νέα χρήματα και όταν έρθουμε στι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε εξασφαλίσουμε μια ρύθμιση η οποία θα δώσει πολύ περισσότερα λεφτά στο μέλλον. Τώρα υπάρχει μια απλή ερώτηση. Την έχετε. Παρακαλώ κύριε Ντεβά, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ που μου δίνει το δικαίωμα να κάνουμε ερώτηση. Και σέβομαι τις γνώσεις του κυρίου Χάουιτ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δουλειά του παρελθόν, οπότε το ερώτημά μου είναι το εξή. Πώ, θεωρείτε τις τις ε, δικές μας υποθέσεις για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία που έχουν μια χριστιανική παράδοση στην Ευρώπη και αναμένεται να το δεχτούν άλλοι πολιτισμοί η θρησκείες, η έλλειψη θρησκειες να καταλάβουν ακριβώς το τι λέμε χωρίς να φαίνεται πως επιβάλλουμε νεοαπικιακές ιδέες. Πώς θεωρητικό αυτό. Ευχαριστώ. 30 δευτερόλεπτα δει, κύριε Χαουίτ. 30 δευτερόλεπτα για αυτή την ερώτηση είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά η απάντηση είναι πω όλοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να ξέρουν πω η ελευθερία σκέψη και θρησκεία είναι θεμελιώδη δικαίωμα για όλα τα έθνη, τι χώρε του ανθρώπου και του λάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Μόλτσερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, η αναπτυξιακή βοήθεια δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και συχνά βλάπτει κιόλα γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα προβλήματα της κάθε χώρας. Δεν υπάρχει συνέχεια και συντονισμός. Το αν θα αλλάξει κάτι ένα πανευρωπαϊκό μέσο είναι κάτι για το οποίο αμφιβάλλω γιατί βεβαίω δεν υπάρχει μια συνεκτική στάση αν δίνουμε σε μικροαγρότες της ε, Αφρικής ε, λεφτά και μετά τους καταστρέφουμε με την επιδοτούμενη γεωργική πολιτική μας απλά σπαταλάμε δισεκατομμύρια Επίσης η κινέζικη αναπτυξιακή βοήθεια με την οποία όπως ξέρετε εξασφαλίζει το Πεκίνο πρώτες ύλε ανταγωνίζεται την δική μας πολιτική και είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Επίσης, τα αναπτυξιακά χρήματα βεβαίω ε, θα πρέπει να αποτελέσουν όρο, θα πρέπει να έχουν ως όρο την επανεισδοχή προσφύγων. Ευχαριστώ κύριο Μπέρμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το κοινοβούλιο αυτό ζητάει αυτό το οποίο ζητάει κάθε κοινοβούλιο στον κόσμο, δημοκρατικό έλεγχο και λόγο στην διεξαγωγή της πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πρότυπο παγκοσμίω και γι' αυτό η συνθήκη τη Λισαβόνα απετέλεσε σημείο πρόοδου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η μεγάλη πλειοψηφία εδώ πέρα δεν είναι ικανοποιημένη από τι προσπάθειε Κοινοβουλίου και Κομισιόν να μειώσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε σχέση με αυτά τα οποία λέει η συνθήκη. Δεν θέλουμε να διαχειριστούμε όλε τι λεπτομέρειε, απλά θέλουμε να έχουμε επιρροή και έλεγχο στρατηγικέ επιλογέ και την ουσία τη πολιτική Σε άλλε χώρε ο κόσμο βγαίνει στου δρόμου για να ζητήσει αυτό τον έλεγχο και πρέπει βεβαίω να του στηρίξουμε. Αλλά ο αγώνα για τη δημοκρατία γίνεται και με δύσκολε διαπραγματεύσει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πως αυτοί οι οποίοι ζητάνε μέγιστο δημοκρατικό έλεγχο έχουν δίκιο είτε στο Κάιρο τη Τίνιδα είτε στι Βρυξέλλες. Ευχαριστώ κύριο Γκρίφιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μία νεαρή γυναίκα στην εκλογική μου περιφέρεια όπω κάθε μέρα μου είπε ότι γύρισε στο σπίτι αφού πήγε τα παιδιά τη στο σχολείο. Η Τζέννη τα πήγαινε τα παιδιά με το αυτοκίνητό τη, αλλά τώρα δεν έχει λεφτά να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό τη. Και δεν έχει λεφτά να πάει να αγοράσει και τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ στο Μάντσεστερ. Πεινάει η, η Τζέννη δεν έχει αρκετά λεφτά για να πάρει ψωμί και τρόφιμα. Εμείς συζητάμε συνέχεια για χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία σημαίνουν 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ χρημάτων φορολογουμένων για την προώθηση της δημοκρατίας και των ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων στον τρίτο κόσμο όλο και περισσότερο μειώνεται η εποπτεία και η εξουσία που έχουν τα κράτη-μέλη, όσο η Κομισιόν απορροφά όλο και περισσότερα χρήματα του Βρετανού φορολογούμενου. Τι σπατάλει αυτό και τι υποκρισία να δίνουμε λεφτά στην Αφρική όταν η Τζέννη και χιλιάδε τόσε άλλε γυναίκε στην Αγγλία δεν έχουν να φάνε. Ο κύριο Κούτε, ένα λεπτό έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και μου. Δεν θα συζητούσαμε αυτό το θέμα εάν ε, κάποιες ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είχαν ζητήσει διατάξεις μέσα στη συνθήκη για τις πρώην απικίες τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αναδειχθεί σε μια πολιτική που βασίζεται στην εκρίζωση της φτώχειας, στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εργατικού δικαίου, της εξεπρεπούς εργασίας ε, και ούτω καθεξής. Οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι πλέον στρατηγική εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και άρα η συνεργασία έχει κέρια σημασία διότι διευκολύνει γενικότερα την οικονομική συνεργασία των χωρών ε, και γι' αυτό θα ήταν καλό να τονώσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις και να ενισχύσουμε τις εταιρικέ σχέσεις ανάμεσα στους ε, δημοσίους φορείς και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, ευχαριστώ, κύριε Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην άμεση γειτονιά μας φεύγουν οι δικτάτορες και αυτό είναι θετικό. Και επειδή οι δικοί μας ε, οι εκπρόσωποι δεν είναι σε θέση ή δεν έχουν τη θέληση να υποστηρίξουν αυτούς που ζητάνε τη δημοκρατία, είναι τουλάχιστον καλό να μην μιλάμε μόνο, αλλά να κάνουμε και καμία πράξη και να βοηθήσουμε. Και αυτή η βοήθεια πρέπει να συνδέεται με τις αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των βασικών συνθήκων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να βοηθάει μόνο, αλλά να ενισχύει αυτές τις αξίες που μας έκαναν ισχυρούς. Και είναι σαφές για μένα πως αυτή η βοήθεια θα πρέπει να ρυθμίζεται και να ελέγχεται από ένα δημοκρατικό κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να δρά η Ένωση και να τα ελέγχουν αυτά οι υπάλληλοι. Όχι. Πρέπει να έχει το δικαίωμα το κοινοβούλιο να κάνει αυτά τα οποία έχει ως δημοκρατικό κοινοβούλιο, δηλαδή να λαμβάνει τελική απόφαση. Ευχαριστώ κύριε Λάιχθριντ. Τώρα περνάμε στην διαδικασία KHDI. Ως πρώτος έχει τον λόγο. Πρώτη η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει ίσα δικαιώματα με το Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση των ε, στρατηγικών σχεδίων για την ε, απορρόφηση των ε, κονδυλίων από τα μέσα αναπτυξιακής βοήθειας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι διαλλακτική η Ευρωπαϊκή Ένωση να επισπεύσει τη, λειτουργία, τη θέση λειτουργία αυτών των μηχανισμών που μας επιτρέπουν να συνεργαζόμαστε με τις χώρες και Οφείλουμε να έχουμε ρεαλιστική προσέγγιση στις σχέσεις μας με αυτές τις χώρες εταίρους. Κρίνω επίσης ε, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μέσα ε, στην Τουρκία, στο Τουρκμενιστάν ε, που μπορούν να μας προσφέρουν ενεργειακούς πόρους μέσα από στρατηγικά σχέδια όπως ο αγωγός Ναμπούκο. Θα ήθελα τώρα να παραπέμψω στην κοινή δήλωση του Πρωθυπουργού της Ρωμανίας και του Προέδρου του Τουρκμενιστάν για την εταιρική σχέση σχετικά με την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου ε, και την μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Το ίδιο ισχύει και για την Αρμενία και τη συνεργασία που είχε με το Ιράκ για την ανοικοδόμηση της χώρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τα μέσα αυτά που είναι αφιερωμένα στην ανάπτυξη των χωρών του τρίτου κόσμου μέσω κάποιων διάβλων τα λεφτά πηγαίνουν σε εταιρείε και μονοπόλια στις ε, δικές μας χώρες. Θεωρώ πως ε, το βασικό μέρος ε, των χρημάτων αυτών θα πρέπει να πηγαίνει, να διατίθεται σύμφωνα με τα έργα εκείνα τα οποία θέλουμε να στηρίξουμε. Πολλοί υπουργοί μου λένε πως συχνά χρηματοδοτούμε δικτατορίες και καθιστώτα τα οποία κάθε άλλο παρά δημοκρατικά είναι. Όταν μιλάμε λοιπόν για ανάπτυξη των πιο φτωχών ε, χωρών πρέπει να διαθέσουμε τις ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βάγκελ, περνάμε τώρα ξανά στην Επιτροπή. Ο Επίτροπος, ο κύριος θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις ε, συνεισφορές σας στη συζήτηση Ελπίζει η Κομισιόν ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για τα σημαντικά αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρέπει όμως να είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε πλήρως αυτά τα εργαλεία στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να είναι όμοιρος η δράση στον τομέα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από διαφορές μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει εμείς να χάσουμε λοιπόν τη σημασία που μπορούμε να έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό η Κομισιόν είναι έτοιμη να βοηθήσει τα δύο αυτά θεσμικά όργανα για να ξεπεράσουν τις διαφορές τους. Τα τωρινά εργαλεία τα οποία ισχύουν μέχρι το 2013, δηλαδή για τα επόμενα δύο χρόνια, όταν όλα τα μέτρα τα οποία θεωρούνται ότι είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του του προπολογισμού εμπλέκονται στη διαδικασία τη επιτροπολογία. Τα έγγραφα στρατηγική είναι τεχνικού έγγραφα και επομένω λόγω τη φύση του δεν μπορούν να έχουν το χαρακτήρα δεσμευτικών νομικών πράξεων. Τα τωρινά εργαλεία έχουν δύο ακόμα χρόνια μέχρι την εκπνοή του και παραμένουν ελάχιστα μονάχα στρατηγικά έγγραφα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν. Η Κομισιόν <clears throat> θεωρεί ότι μια αλλαγή αυτού του συστήματο τώρα θα απαιτήσει πολλές αλλαγές στα εργαλεία αυτά που θα χρειαστεί πολύ χρόνο και θα είναι αντιπαραγωγικό για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν εμπλέκει ήδη πλήρω στο Κοινοβούλιο στην ε, παρακολούθηση των δράσεων αυτών υπέρ τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει λοιπόν εκτεταμένα δικαιώματα ελέγχου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τα νέα εργαλεία είναι πολύ νωρί να πούμε, είναι πρόημο να πούμε τι ακριβώ χαρακτήρα θα έχουν γιατί χρειάζεται μια διαβούλευση με όλου του εμπλεκομένους βάσει τη προτάσεω τη Κομισιόν. Εφόσον τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 290 τη Συνθήκης Λισαβόνα. την χάνουν πλήρου σεβασμού, έχουμε την επιλογή να υπάρξει και προσφυγή σε πράξεις κατ' και στη νέα περίοδο προγραμματισμού. Η Κομισιόν δεν έχει ακόμα σταθμισμένη άποψη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Λέει Πρόεδρος, οι εισηγητές τώρα έχουν την ευκαιρία να λάβουν και πάλι το λόγο. Ξεκινά πρώτα ο κύριος Γκέρντς. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν για τα μέσα συνεργασίας και αναπτυξιακής βοήθειας ε, που είναι και το αντικείμενο της έκθεσής μου. Ο Έλμαρ Μπρόκ νομίζω ε, εκφράστηκε πολύ εύστοχα, ε, εξέφρασε αυτό που θέλουμε. Δεν θέλουμε να γυρνάμε γύρω-γύρω και να μην είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά ούτε και θέλουμε να δώσουμε στο εκτελεστικό σκέλος της Ένωσης μια επιταγή εν λευκό για να εφαρμόσει διατάξεις που ε, ουδόλως υπάγονται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μια ισορροπημένη λύση χρειαζόμαστε ούτως ώστε να χρησιμοποιούμε σωστά τα στρατηγικά σχέδια και τις πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση συνέχεια. Μόνο αυτό διεκδικούμε, μόνο αυτό αξιώνουμε. Ε, ευχαριστώ και όλους όσοι ήταν ε, επικριτικοί και εξέφρασαν ε, σκεπτικισμό για την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Βέβαια αναφέρονται ε, στους φορολογουμένους ε, και θέλουν να μην έχει κανένα έρισμα η αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Κοιτάξτε, οι φορολογούμενοι χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό που χρηματοδοτεί δράσεις αλληλεγγύης προς τους μη έχοντες. Αυτό ε, καθίσταται δυνατό χάρη στη συμβολή των φορολογουμένων που από τη χώρα τους συνδράμουν στη διαδικασία και Προφανώς θέλουμε να ε, προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των απόρων, των μη εχόντων. Θα ήθελα να παραπέμψω τους ε, επικριτικούς συναδέλφους ε, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ. Θα διαπιστώσουν εκεί ότι όσοι κάνουν τα περισσότερα στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας και της εξωτερικής αλληλεγγύης είναι οι ίδιοι που δαπανούν περισσότερα για την εσωτερική αλληλεγγύη στη χώρα τους. Ε, δεν υπάρχει αντινομία, δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην ε, εγχώρια και την εξωτερική αλληλεγγύη και όσοι θέλουν να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι τα κονδύλια που δαπανώνται για την εξωτερική αλληλεγγύη ε, ε, ε, ισοδυναμούν με διασπάθηση του δημοσίου χρήματος να πάμε να διαβάσουν το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ. Παρακαλώ η κυρία Λοχπίλτερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ πως έγινε σαφές ε, με τη συζήτηση για τις ε, κατεξοδότητες πράξεις το γιατί τις θέμε. Δεν θέμε να κάνουμε μικροδιαχείριση, θέλουμε να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις πληροφορημένοι και να προλάβουμε λάθος εξελίξεις ή να τις διορθώσουμε αν αυτό είναι απαραίτητο. Και όταν εκπροσωπούμε το Κοινοβούλιο προς τα έξω, π.χ. με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επηρεάζονται όταν στο μέλλον ε, δεν θα υπάρχει καμία χρηματοδότηση για τα έργα, τότε βλέπω πως συμφωνούν και αντιλαμβάνονται τη θέση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή δεν είναι πως δεν θα αντιλαμβανόταν μια λογική τοποθέτηση στο Κοινοβούλιο. Επίσης, για την κριτική που ασκήθηκε ότι ξοδεύονται πάρα πολλά λεφτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Εγώ πρέπει να διαπιστώσω το αντίθετο. Εάν δούμε το μέσο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, διαπιστώνουμε, υπάρχει από το 2004 μόλις, πως έχει σχετικά λίγα λεφτά και με αυτά μπορούν να γίνουν αρκετά πράγματα. Βεβαίω, αυτά δεν μπορεί να δίνονται έτσι διακρίτως, πρέπει να δούμε τι έχουν επιτύχει τα διάφορα έργα και σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις έπρεπε να διακοπούν κάποια συγκεκριμένα έργα. Εάν θέλουμε αυτές τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να ζει ο κόσμος ελεύθερος και ελεύθερος από ανάγκη, τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε προς τα εμπρός. Και άρα αυτό το μέσο είναι πάρα πολύ καλή συμπλήρωση πολιτικής που ασκούμε και ζητάμε από άλλες χώρες. Οπότε δεν είναι πάρα πολύ Δεν είναι πάρα πολλά τα λεφτά, αντιθέτως πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη. Ευχαριστώ κυρία Λοχμπίλερ. Τώρα η κυρία Γκάλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο, καθώς και τον κύριο Επίτροπο για τις ε, παρατηρήσεις τους. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με υποστήριξαν. Ο κύριος Μπρόκ είπε κάτι το οποίο ήταν πολύ σαφές, ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ νομοθετικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη των δύο. Αλλά τόσο <clears throat> οι εισηγητέ, όπω και πολλοί βουλευτέ, τόνισαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρόλα αυτά θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ενό δικαιώματο συναπόφαση και συνδιαβούλευση για την ε, χάραξη τη στρατηγική σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν εκεί που είναι πιο απαραίτητα. Σε σχέση λοιπόν με τη χρήση των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων, εγώ δεν πιστεύω ότι ο φορολογούμενος θέτει αναφιβόλο τη σημασία αυτών των εργαλείων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, πολλές φορές την ζωή ακόμα των ανθρώπων υποστηρίζουν αυτά τα εργαλεία. Εγώ νομίζω ότι οι φορολογούμενοι κατανοούν την αξία αυτών των εργαλείων και τα υποστηρίζουν. Και θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει <clears throat> να χρησιμοποιήσει τις νέες αρμοδιότητες που το έχει δώσει η Συνθήκη της Λισαβόνας και θα χαρώ πάρα πολύ για αυτό το λόγο αν το Συμβούλιο και η Κομισιόν εργαστούν για να υπάρξει μια πραγματικά θετική συμβαστική λύση για όλους που θα μας δώσει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και αυτό απαιτεί τη συνεργασία και των τριών μεγάλων θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μίτσελ έχει το λόγο, ο οποίος θα τοποθετηθεί με μία δήλωση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, βλέπω πως μου δίνετε λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί δεν μπόρεσα να μιλήσω στην αρχή. Ε, με συγχωρείτε, είχα κολλήσει την κίνηση. Ε, συνάδελφοι ανέφεραν την κατάσταση σε σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν λειτουργούσαν η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη-μέλη μας, τότε δεν θα πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο με μια φέτα ψωμί και λίγη μαρμελάδα. Εάν αυτή είναι η κατάσταση στη Βρετανία και σε άλλα κράτη-μέλη, τότε πρέπει να διασφαλίσουν τα κράτη-μέλη πω δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το θέμα μα εδώ πέρα. Όχι μόνο η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 22.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα κάθε μέρα σε μικρή απόσταση με το αεροπλάνο από αυτό εδώ το κτίριο. 22.000. Τα καλά νέα είναι πως ήταν 34.000 αυτός ο αριθμός. Φροντίσαμε να κατεβάσουμε αυτόν τον αριθμό λόγω της χρηματοδότησης ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ας μην βάζουμε αυτούς τους ανθρώπους έναντι το να πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά στο σχολείο με τα πόδια. Κάτι για το οποίο επίσης ε, λυπάμαι. Το θέμα αυτό αφορά την εφαρμογή ή της πράξεις κατεξιοδότησης, στην περίπτωση στην οποία μιλάμε για νομοθεσία. Εγώ προτείνω να μείνουμε στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και άρα να πούμε πως θα επαναφέρουμε όλες τις τροπολογίες μας καθώς το ζήτημα είναι κρίσιμο για το μέλλον των διοργανικών σχέσεων στον τομέα των εξωτερικών δράσεων. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου δεν αφορούν την ουσία του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας ή οποιοδήποτε άλλο μέσου, αλλά την εφαρμογή του ρόλου του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα δημοκρατικά προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως προβλέπονται οι συνθήκες της Λισαβόνας. είναι νομοθέτες πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε όπως και το Συμβούλιο η υιοθέτηση και εκτέλεση στρατηγικών αποφάσεων για τη διάθεση αναπτυξιακής βοήθειας. Πώς, από και πώς. Σε τακτικούς όρους διασφαλίζουν τροπολογίες πως κάποια σχέδια οι αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την Κομισιόν αναγνωρίζονται ως πράξεις κατά εξιοδότηση όπως ορίζονται στο άρθρο 209 της Συνθήκης. Έτσι, οι δύο συνομοθέτες θα μπορέσουν να έχουν αντιρρήσεις σε σχέδια αποφάσεων που δεν συμφωνούν με τον νόμο. Ε, με αυτό το βέτο θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του Κοινοβουλίου όταν προγραμματίζει κοινοτική βοήθεια η Δεν μιλάμε για διαχείριση, όπως είπαν οι συνάδελφοι, μεμονωμένων προγραμμάτων. Τροπολογίες θα διασφαλίσουν πως οι νομοθέτες θα έχουν έλεγχο στις στρατηγικές αποφάσεις για τις προτεραιότητες και τους τομείς. Όλες οι τροπολογίες είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην πρώτη ανάγνωση στη θέση του Κοινοβουλίου που είχαν υιοθετηθεί την 21 Οκτωβρίου που μας πέρασε. Αλλά τις απέρριψε όλες το Συμβούλιο χωρίς να προτείνει καμία εναλλακτική λύση που θα ικανοποιούσε τις απαιτήσει του Κοινοβουλίου. Είναι ατυχές πως στο ένα έτος σχεδόν που πέρασε από την πρώτη συζήτηση του φακέλου στην Επιτροπή, οι δύο οργανικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν σημειώσει πρόοδο και σας διαβεβαιώ πως προσπαθήσαμε πάρα πολύ στις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, οι οποίες ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2010. Είχαμε τρεις διαλόγους και πολλές τεχνικές συναντήσεις, αλλά δεν είχε υπάρξει κάποια προσέγγιση μόνο προς το τέλος του περασμένου έτους ε, έκαναν μια συμβαστική πρόταση οι διαπραγματευτές της Κομισιόν αμέσως ανταπάντησε το Κοινοβούλιο αλλά δεν πήγε αυτή η θέση επισήμως στην συνεδρίαση του Συμβουλίου παρά τη σκληρή γραμμή του Συμβουλίου με την οποία συμφωνεί και η Κομισιόν και λυπούμε γιατί δεν είναι η θεσμική τους θέση να το κάνουν. Εμείς επιμένουμε στη θέση μας. Νομικά τα επιχείρηματα μας στέκουν, τα στρατηγικά έγγραφα των ε, πολιετών προγραμμάτων ε, εκπληρώνουν τα κριτήρια για την διαδικασία πράξεων κατεξιοδότηση. Τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 290 είναι υποχρεωτικά. Εάν πληρούνται πρέπει Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να έχουν δικαίωμα βέτο. Δεν είναι θέμα εδώ πέρα πολιτικής συμφωνίας, καθώς ε, αυτά αναφέρει η συνθήκη. Είναι νομική μας υποχρέωση. Έχουμε την πλήρη στήριξη της διάσκεψης των Προέδρων που αποφάσισε σε δύο συνεδριάσεις και μάλιστα αυτό τον μήνα πως σε όλες τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να επιμένουμε στην διαδικασία αυτή για αποφάσεις που αφορούν προτεραιότητες, κατανομές και γενικούς στόχους. Επίσης έχουμε κοινή γραμμή μεταξύ των επιτροπών, οι επιτροπές ανάπτυξης και εξωτερικών υποθέσεων, πως και οι υπόλοιποι εισηγητές, όπως ξέρετε, έχουν υιοθετήσει την ίδια στάση. Όλες οι τροπολογίες θα πρέπει να επανεισαχθούν. Η θέση μας είναι απλή και σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει η διάσκεψη των Πρόεδρων δεν θα ε, μας διαχωρίσετε ούτε θα αγνοήσετε τον ρόλο μας ως νομοθέτη. Είμαι επίσης πεπισμένος πως έτσι θα ωφεληθούν και οι δικαιούχοι. Το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει πολύ πιο αποτελεσματικά τον ρόλο του για να φροντίσει να πηγαίνουν τα λεφτά εκεί όπου ορίζει η συνθήκη για την αναπτυξιακή βοήθεια της Ένωσης. Η μείωση και η εξάλληψη της φτώχειας 22, δεν χρειάζεται να πεθάνουν 22.000 παιδιά κάθε μέρα. Απαιτούμε λοιπόν να έχουμε κι εμείς λόγο σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μίτσελ. Είχατε προφανώς περισσότερο χρόνο γιατί δεν ομιλήσατε στην αρχή της ε, συζήτησης. Έχετε μια μπλε κάρτα τώρα. Ο κύριος Ντέβα θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα. κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον έντιμο συνάδελφο και φίλο μου κύριο Μίτσελ κατά πόσο θα συμφωνούσε μαζί μου ότι το 2005 το Κοινοβούλιο ουσιαστικά άφησε να φύγουν από τα χέρια του 14 περιοχές συναπόφασης για αυτά τα εργαλεία χρηματοδοτικά. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τα πάρουμε πίσω. Γιατί εμείς όχι μόνο <clears throat> χάσαμε την ευκαιρία να ξέρουμε τι κάνει η Κομισιόν, Χάσαμε τη διαδικασία λογοδοσίας για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μίτσελ λοιπόν να συμφωνεί σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε παρακαλώ κύριε Μίτσελ. Συμφωνώ με τον κύριο Ντίβα ότι χάσαμε εχωρίσαμε κάποια από τα δικαιώματά μας. Ήμουνα τότε εισηγητή για το Εργαλείο Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Δύο χρόνια χρειάστηκε για να συμφωνήσουμε, γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε μερικά από τα βασικά δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Θέλαμε, χρειάστηκε όμως να κάνουμε συμβασμού στο τέλος. Και υπήρξε μια θεσμική, διαθεσμική συμφωνία με τη Κομισιόν και το Συμβούλιο που είχε σαν αποτέλεσμα εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης να έχουμε δικαιώματα εποπτείας για το Εργαλείο Ανάπτυξης και Δημοκρατίας και αυτό ήταν το πνεύμα τη συμφωνία αυτή που θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Ω τελευταίο ομιλητή, ο κύριο Σόλτ, για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Δεχούχτ, έχετε δίκιο ότι είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε αυτό το πράγμα. Ελπίζω ότι θα μπορέσει στη δεύτερη ανάγνωση να επιτευχθεί μία συμφωνία. Και πρέπει επίσης να θέσουμε και το ερώτημα. Γιατί μια αρχή η οποία είναι σαφώς εδρεωμένη στη συνθήκη και έχει νομικό χαρακτήρα δεν γίνεται σεβαστή. Τόνισε ο κύριος Μπροκ πολύ σωστά ότι εδώ πρόκειται για να έχει το Κοινοβούλιο να διαβουλεύεται και να παίζει ρόλο στην, στον καθορισμό των στόχων. Στα πολιτή σχέδια της Κομισιόν για το DCI, για το εργαλείο αυτό της ανάπτυξης, Υπάρχει μια μνήα της στρατηγικής Global Europe και την συνδέει η Κομισιόν με την ε, ε, χρηματοοικονομική κρίση στην Ευρώπη και τονίζει ότι είναι σημαντικό να μπορέσει να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία διότι έχει προβλήματα να διεισδύσει σε διάφορες αγορές. Εδώ σας λέω και πάλι ότι δεν ήταν αυτός ο στόχος για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το εργαλείο από τον νομοθέτη και κατά την άποψή μας αυτό θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τη συνεργασία και όχι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιεί η Κομισιόν κατά το δοχκούν. Για μας οι χώρες της ε, Νοτιοανατολικής Ασίας δεν είναι η μόνη εταίρη της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είπε η Κομισιόν πρέπει επίσης να συνεργαστούμε και με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και όχι μόνο να τις βλέπουμε σαν πηγές φυσικού αερίου και φυσικά για τις χώρες του Μαγκρέπ έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και να συνεργαστούμε μαζί τους. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων κρατών με διαδικασία η οποία θα εμπλέκει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς το συμφέρον των πολιτών μας σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόλτς. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει κλείσει η κοινή συζήτηση για τα θέματα αυτά των χρηματοδοτικών εργαλείων και σήμερα στις 11.30 θα γίνει η ψηφοφορία για τα θέματα αυτά.